Βλέπετε έγινε αλλαγή φρουράς λέει ο πρόεδρος. Και συνεχίζει στα τσεχικά. Θα προχωρήσουμε στη δήλωση της ε, υπάτης ε, ε, προσώπου για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Κυρία Άστον έχει το λόγο. Παρακαλώ. Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, σας ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ διότι μου δίνεται η ευκαιρία στη σημερινή συζήτηση να τοποθετηθώ για την ενευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και με ενδιαφέρει πολύ η άποψη των αξιότιμων βουλευτών. Εγώ πιστεύω ότι ε, είναι επίγουσα η ανάγκη να σημειωθεί πρόοδο στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Όπω λέγαμε και στο Κοινοβούλιο σήμερα το πρωί, βλέπουμε τι ραγδαίε ιστορικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Τινησία και στην Αίγυπτο και ε, την ε, βία στο, στη Λιβύη, στο Μάν, στο Μπαχρέιν και σε άλλε χώρε. κλειδονίζεται ολόκληρη η περιοχή και παρόλα αυτά κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν είναι η ώρα, η κατάλληλη στιγμή να εστιάσουμε την προσοχή μα στην ειρηνευτική διαδικασία τη Μέση Ανατολή. Εγώ πιστεύω ότι ισχύει το αντίθετο. Αυτή ακριβώ τη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να τερματίσουμε αυτήν την σύραξη. Έτσι θα συμβάλλουμε ε, στην σταθερότητα ε, και στην ειρήνη στην περιοχή. Αυτό το μήνυμα πέρασα ε, όταν μετέβηνε επιτόπου τον Ιανουάριο και τον Φεβρουαρίο συζήτησα με τον πρόεδρο Αμπά και τον πρωθυπουργό Νετανιάχου για την ειρήνη ε, ε, και των δύο λαών θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία. Επίσης πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Ε, το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στα συμπεράσματά του στο Δεκέμβριο τοποθετήθηκε για αυτό το θέμα. Η μόνη βιώσιμη λύση είναι μια διαπραγμάτευση και <clears throat> που θα οδηγεί σε μια λύση για τα δύο κράτη. Για να υπάρξει ειρήνη θα πρέπει να λυθεί το θέμα της μελλοντική πρωτεύουσα Ιερουσαλήμ και για τα δύο κράτη. Ε, για την, ε, ε, θα πρέπει να υπάρχει ένα κυριαρχό ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος που θα συμβιώνει ειρηνικά με το Ισραήλ. Γνωρίζετε τη θέση μας για τους επικισμούς, είναι παράνομοι, συνιστούν πρόσκομα για την ειρήνη και απειλούν την εξέβρεση λύσης για δύο διαφορετικά κυρίαρχα κράτη. Τον, στο Μόναχο 5 Φεβρουαρίου τοποθετηθήκαμε ε, ε, στο πλευρό των, ε, του, του κουαρτέτου και συμφωνήσαμε με τα Ηνωμένα Έθνη, με τη ΣΥΠΑ και την ε, Ρωσία για ένα φιλόδοξο σχέδιο. Ε, συναντηθήκαμε την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Προείδρευσε ο κύριος ε, Σμιτ, πολιτικός διευθυντής της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και για πρώτη φορά ακούστηκαν και οι διαπραγματευτές από την Παλαιστίνη και την ερχόμενη εβδομάδα θα ακούσουμε τους Ισραηλινούς διαπραγματευτές ε, τώρα προετοιμάζουμε την επόμενη βασική δίσκεψη όπου ο Βαν Κιμούν, ο Βολάνβεροφ, η κυρία Κλίντον και ε, εγώ θα συμμετάσχουμε ούτως ώστε να βρούμε μια λύση βιώσιμη. Το τονίζω, αυτό χρειαζόμαστε και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό ε, να τοποθετηθούμε διότι εμείς δίνουμε σημαντική βοήθεια στους Παλαιστινίους και θέλουμε να συνεχίσουμε να τους υποστηρίζουμε για την ανοικοδόμηση του κράτους και την εφαρμογή του σχεδίου. Θέλουμε να στηρίξουμε πολιτικά και οικονομικά. Έχουμε ήδη εγκρίνει ε, τα πρώτα 100 εκατομμύρια ευρώ από τα 300 που θα δοθούν συνολικά ε, και θα εκταμιευτούν το Μάρτιο 2011. Ε, τώρα για την συγκρότηση των δημοκρατικών θεσμών είναι ένα απαραίτητο βήμα ούτως ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν ως κυρίαρχα κράτη και είναι κέρια σημασία και για την Παλαιστίνη και για ε, το Ισραήλ για να έχουμε μία βιώσιμη λύση δύο ξεχωριστών ε, κρατών. Ξέρετε ότι πήγα στην ε, Λωρίδα της Γάζας, συναντήθηκα με κοινωνικούς εταίρους, συναντήθηκα και με πολλά παιδιά και προτείναμε ένα συνολικό πακέτο βοήθειας για την υποδομή, τον τεχνικό εξοπλισμό και την εκπαίδευση. Το πέρασμα του Κάρι Σαλάμ είναι πάρα πολύ σημαντικό για να διακινούνται τα αγαθά, ε, επιτρέπουμε έτσι τις εξαγωγές ε, και ε, θα επέλθει η οικονομική ανάκαμψη. Επίσης, ζήτησα να υπάρξουν μεγαλύτερες ευκαιρίες για τον τόπιο πληθυσμό, να έχουν θέσεις εργασίας, να εξασφαλίσουμε την οικονομική ανάπτυξη και κυρίως να φροντίσουμε τα παιδιά. συνεχίζω λοιπόν να απευθύνω την έκκληση για να απελευθερωθεί ο Μπίρες Σαλίντε και επίσης στην, στο Συμβούλιο Σύνδεσης ad hoc, στη στις 30 Απριλίου θα ε, συζητήσουμε και το θέμα της διάσκεψης αδωρητών για τον Ιούνιο που ενδεχομένως να διεξαχθεί. Ε, κάναμε πάντως στο Συμβούλιο Σύνδεσης ε, στις 22 Φεβρουαρίου μια επικοδημοτικότατη ανταλλαγή απόψεων. Συζητήσαμε την ενευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και άλλα περιφερειακά ζητήματα και κυρίως φυσικά τις δραχτέ αλλαγές που σημειώνονται στην περιοχή. Με, μεταξύ των θεμάτων που συζητήσαμε είναι οι διμερείς μας σχέσεις, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την μελλοντική μας συνεργασία συνεργασία βάσει ε, του τωρινού σχεδίου δράση ε, και δεδομένου του ότι επιθυμούμε όλοι να εξευρεθεί μια βιώσιμη λύση. Επίση, καλωσορίζω την βούληση του Ισραήλ ε, για την απόφαση του για την αποστολή αύριο. Επίση, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αρχίσουν οι άμεσε επαφέ, οι εκ του σύνεγγυ συνομιλίε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και για του δύο λαού και για τα δύο κράτη. Ο Πρωθυπουργό Νετανιά Νετανιάχου έχει ρόλο κλειδί για να προχωρήσουν τώρα οι διαπραγματεύσει αξιότιμοι βουλευτέ. Θα ήθελα να ακούσω τι απόψει σα με μεγάλο ενδιαφέρον και θα διακόψω τώρα. Απλώ κλείνοντα, θα σα πω ότι κατά τη γνώμη μου όλοι επιθυμούν εδώ μέσα να λήξει επιτέλου η σύραξη και να βρούνε ε, οι δύο πλευρέ σε μία λύση και για το λαό τη Παλαιστίνη και για το λαό του Ισραήλ και για να ενισχύσουμε την σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή. Και απευθύνω θερμή έκκληση προ όλου, ώστε αυτό να συμβεί σύντομα. Σας ευχαριστούμε κυρία Άστον. Ε, θα ήθελα να ακούσουμε τώρα τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Ε, εξ ονόματος του ΕΛΚΟ, κύριο Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ κύριε Πατηγβόσοπη και αντιπρόεδρε. Αξιότιμη συναδέλφα, πολύ σωστά κύριε Άστον το είπατε. Η κατάσταση όσον αφορά την νότια όχθη της Μεσογείου ε, μας αποστρέφει την προσοχή από τη Μέση Ανατολή και από την ενευτική διαδικασία και επομένως εδώ και 30 χρόνια είχε αρχίσει αυτή η διαδρομή και τώρα βρισκόμαστε ε, σε μια κατάσταση αποτελματωμένη. Πήγατε και θα πρέπει να προβληματιστούμε όσον αφορά την επίσκεψή σας. Και τώρα έχω κάποιες ερωτήσεις σχετικά για να μου πείτε τη γνώμη σας. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε τα θέματα τα σχετικά με τις υπάρχουσες δυσκολίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας δυσκολίες όσον αφορά ένα επιπλέον ψήφισμα για την περίπτωση κάποιας ε, ζώνης απαγόρευσης υπερπτήσεων. Θα ήθελα εσείς τώρα να μας αξιολογήσετε σε ποιο βαθμό αυτό θα επηρεάσει την ενευτική διαδικασία και την αξιοπιστία μας. Αυτό το βέτο, αυτή η άρνηση κυρία σε σχέση με την καταδίκη τη σχετική με τα γεγονότα για τους επικισμούς στην Παλαιστίνη. Άρα, τι θα πρέπει να γίνει θεωρείτε ώστε να ενεργοποιηθεί ο Ομπάμα να επέμβει. Επίσης τι λέτε όσον αφορά την Παλαιστίνη που θέλει να κάνει κοινοβουλευτικές και προεδρικές εκλογές πριν το Σεπτέμβριο και ε, την αρνητική πρόθεση της, ε, της Χαμάς για αυτές τις ερωτές. Επίσης πώς αξιολογείται τον Παλαιστίνιο ηγέτη που κατηγορήθηκε μέσω του Wikileaks όσον αφορά ε, την Παλαιστινιακή Αρχή ε, και αυτές οι κατηγορίες πόσο έχουν επηρεάσει την Παλαιστίνη και το Ισραήλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι βλέπω μία κάρτα μπλε από τον κύριο Κάλαχη. Θέλετε το λόγο. Κύριε Σαλαφράγκα, ε, δέχεστε την επερώτηση. Ναι, ναι. Έχετε το λόγο. Κυρία Άστον. Όχι, όχι, όχι, για την κυρία Άστον είναι η ερώτηση, αλλά δεν με βλέπετε. Και ε, ε, ήλξε την προσοχή σας όταν δώσατε το λόγο στις πολιτικές ομάδες. Καλά, θα σας δώσω την ε, ευκαιρία να μιλήσετε όταν κάνουμε το διά. Σας παρακαλώ Πρόεδρε, πρέπει να κοιτάτε και από εδώ και από αυτή την πτέρυγα του ημικυκλίου. Δεν γίνεται αλλιώ. Είναι αδύνατο να σας ελκύσει προσοχή. Πέντε λεφτά κούναγα την μπλε κάρτα. Έχετε. Για την μπλε κάρτα για τους συναδέλφους, όχι για την υπάτη εκπρόσωπο. Τέλος πάντων, Κατά την διάρκεια των μονολέπτων ομιλιών θα σας δώσω την, ε, τον, τον λόγο. Για δύο λεπτά τώρα η κυρία Ντεκάιζε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Άστον. Καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας συζητούμε για την ε, φανταστική ελπίδα που γεννάται από τις εξεγέρεσεις ε, στη Βόρεια Αφρική. Μας εμπνέει όλους η δημοκρατία και γνωρίζουμε ότι το δικαίωμα του να ζει κανείς ελεύθερο είναι ένα καθολικό δικαίωμα ή τουλάχιστον πρέπει να αναγνωρίζεται καθολικά. Ισχύει αυτό φυσικά και για τους Παλαιστινίους. Την ώρα που μιλάμε, την ώρα που συζητάμε, ε, υπάρχουν πάρα πολλοί Παλαιστινοί νέοι που δεν έχουν κανένα μέλλον, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, δεν μπορούν να ζήσουν, να εργαστούν, δεν έχουν καμία δυνατότητα ε, να εξασφαλίσουν ιατρική περίθαλψη, ούτε καν τρόφιμα ε, πολλές φορές. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση και νομίζω ότι είναι γενικευμένη αυτή η αίσθηση ότι δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι η κατάσταση. Ποια είναι η λογική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Συμφωνία Σύνδεσής της. Μας ε, μιλήσατε γι' αυτό, εγώ τη διάβασα πάρα πολλές φορές τη Συμφωνία. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταγγείλει την παραβίαση αυτού του καθολικού, του διεθνούς δικαίου, ζητώ συγγνώμη, επανειλημμένα, τι γίνεται, χωρίς κανένα αντάλλαγμα ε, ζητάτε θετικά κίνητρα, έτσι τα αποκαλείτε, για τη γεωργία, για την αλία, για το περιβάλλον, για τις αστυνομικές δυνάμεις, για τη δικαστική συνεργασία, για τις μεταφορές, ε, για τη διαστημική συνεργασία, επιστημονική συνεργασία, χωρίς να ζητάτε κανένα αντάλλαγμα, χωρίς ένα αντιστάθισμα. Και όταν συνεδρίασε το κουαρτέτο, τους καλέσατε τους Ισραηλινούς, δεν ήρθαν όμως. Θα ήθελα να σας πω λοιπόν, ε, κυρία Άστον, ότι ε, ναι, αναγνωρίζω ότι καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες, ε, αλλά δεν λειτουργούν αυτά τα θετικά κίνητρα όπως τα ονομάζετε. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχουμε δικαίωμα τη σήμερα ημέρα να ε, απορρίψουμε όλα τα μέσα πίεσης, δεν μιλώ για κυρώσεις, ε, στον τομέα της οικονομίας, συγγνώμη, ο χρόνος σας κυρία Κάιζερ διακόπτει ο Πρόεδρος, έχουμε ένα ολόκληρο φάσμα εργαλείων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ενώ παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο και η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό και είναι πολιτικό το ζήτημα και πρέπει να υποφεληθούμε τη ευκαιρία ε, τώρα που έχουμε τι εξεγέρσει ε, στον αραβικό κόσμο. Σα ευχαριστούμε. Ε, κυρία Ντεκάιζερ, μίλησε εξ ονόματο των σοσιαλιστών. Τώρα η κυρία Νίτ Ούτεμπουργκ από του φιλελευθέρου. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ήπατη εκπρόσωπε, εκ μέρου τη δική μου τη πολιτική ομάδα ξεκινώ λέγοντα ότι συμφωνούμε και επαυξάνουμε ε, με αυτά που είπατε στην αρχή, στην εισαγωγή σα και με του ε, στόχου ε, που θέσατε όσον αφορά στις προσπάθειές σας να επαναφέρετε ζωή σε αυτό που αποκαλείται στάσιμη ειρηνευτική διαδικασία και εμείς πιστεύουμε ότι είναι στάσιμη, πρέπει να αναζωογονηθεί έτσι ώστε να σημειωθεί πρόοδος. Την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε την τιμή να δεχτεί εδώ ε, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ ο οποίος ε, ήρθε για να παρουσιάσει την υπόθεσή του αν μου επιτρέπετε να χαρακτηρίσω με αυτά τα λόγια την ομιλία του. Το θέμα είναι ότι ε, δεν ε, εστίασε σε αυτά που συμβαίνουν ε, στα υποκατοχή Παλαιστινιακά εδάφη, αλλά ε, θέλησε να εστιάσει περισσότερο σε τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού Ισραήλ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως για μας θα ήταν πολύ πιο εύκολο να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση αν είχαμε σοβαρές ενδείξεις ότι το Ισραήλ πράγματι επιθυμεί να δώσει νέα όθηση στην ειρηνευτική διαδικασία. Αλλά φοβάμαι ότι το Ισραήλ πιστεύει ότι οι εξεγέρσεις στις ε, αραβικές χώρες ε, του δίνουν ε, μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών. Φοβάμαι κυρία Ντεκάιζερ ότι αυτό θα είναι ένα τεράστιο πολιτικό λάθος. Το Ισραήλ Αντίθετα θα έπρεπε αυτά που συμβαίνουν σήμερα να τα χρησιμοποιήσει για να επιταχύνει την ειρηνευτική διαδικασία και να επιτύχει την ολοκλήρωση της συμφωνίας το συντομότερο δυνατόν. Η κυρία Άουκεν εκ μέρους των Πρασίνων για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την ε, κυρία Άστον για την παρέμβασή της. Ε, είμαι λίγο απογοητευμένη, οφείλω να ομολογήσω, διότι σε αυτή την ιστορική στιγμή ε, στις διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Παλαιστίνης, γιατί δεν ακούσαμε ούτε μία λέξη για την αναγνώριση της, ε, του Παλαιστινιακού ε, κράτους. Ξέρουμε ότι εξέπνευσαν οι προθεσμίες ε, τον ε, Δεκέμβριο. Ξέρουμε ότι πρέπει να σημειωθούν αλλαγές, αλλά η είπατε εκπρόσωπος μας λέει ότι σημειώνεται πρόδοσμα μα ποια πρόοδος. Ε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας ε, είδαμε με σαφήνεια ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνονται πολλά θετικά βήματα σε επίπεδο όμως δηλώσεων, αερολογίες ε, δηλαδή. Πρέπει να επιστρέψετε στον πλανήτη Γη για να συνειδητοποιήσετε ότι είναι σοβαρή η κατάσταση όπως είπε και η κυρία Ντεκάιζερ προηγουμένως το θέμα είναι ότι υπάρχουν οι πολιτικές διαπραγματεύσεις και οι τεχνικές διαπραγματεύσεις ε, αλλά μην ξεχνάμε ότι συνέχεια εξαπλώνονται οι ε, επικισμοί των ε, Ισραηλινών ενώ εμείς συζητούμε είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση γιατί κανείς δεν μιλάει για την χρησιμοποίηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πληρώνουμε, πληρώνουμε, πληρώνουμε και δεν βλέπουμε τα αποτελέσματα γιατί δεν δίνουμε μια ευκαιρία επιτέλους στους Παλαιστίνιους να οικοδομήσουν ένα κράτος. Σε τι χρησιμεύουν όλα αυτά τα λεφτά. Έχουμε αξιοπιστία ε, πραγματικά είναι ιστορική στιγμή, πρόκειται για μια ιστορική καμπή και πρέπει να δούμε πώς θα δράσουμε, όχι να περιοριζόμαστε σε αυτά τα ευχολόγια ε, και να βοηθήσουμε ε, και τις χώρες ε, της Βόρειας Αφρικής και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επίση και τα μέσα πίεση, τα κονδύλια που δίνουμε σε διάφορες χώρες. σα. ευχαριστούμε κυρία Άουκεν. Τώρα από την πλευρά των συντηρητικών ο κύριο Στίβενσον. Ευχαριστώ πολύ κυρία, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι ανησυχώ σοβαρά όσον αφορά τις εξελίξεις ε, στο Ιράκ. Οι τελευταίες εξεγέρσεις εκεί όπου οι άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους, κυρίως οι νέοι που δεν βρίσκουν δουλειά, βλέπουν μια οικονομία που έχει καταρρεύσει, ε, δεν υπάρχει ασφάλεια, δολοφονίες ε, για θρησκευτικού λόγους. Η εξέγερση κατεστάλλει βία, πάρα πολλοί δολοφονήθηκαν, πολλοί και τραυματίες και τώρα υπάρχουν ενδείξεις ότι το κόμμα που κέρδισε τις εκλογές το Μάρτιο θα αποσυρθεί από την συμμαχία διότι ο, ο Πρωθυπουργό ε, δεν κράτησε τις υποσχέσεις του. Εάν λοιπόν ε, συμβεί αυτό τότε θα είμαστε πάλι στο σημείο, υπαρθμών, στο σημείο 0 όπου τόσο ο Χακίμ όσο και ο Χάσσαρα με την υποστήριξη του Ιράν θα αποσταθεροποιήσουν την κατάσταση όπου το κόμμα που θα έχει κερδίσει τις εκλογές δεν θα ε, μπορεί να βρίσκεται στην κυβέρνηση. Αυτό δεν μπορεί να είναι αποδεκτό έχοντας κατά νου το μέλλον της, Ευρωπαϊκής, της ε, Μέσης Ανατολής. Ο κ. Τρενταφυλλίδης παρακαλώ που θα μιλήσει εκ μέρου της ΕΕ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, παίρνω αφορμή από τις ομιλίες που έχουν εκφωνηθεί σήμερα για να αναφερθώ στη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι στα γεγονότα που συμβαίνουν τριγύρω μας στον αραβικό κόσμο. Μια στάση που συχίζει τη στασιμότητα με τη σταθερότητα. Μια επιλείψιμη στάση γιατί απέτυχε να αφουγκραστεί οι απαιτήσει των λαών της περιοχής για ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη. Κι όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμπεριφερθεί διαφορετικά, σωστά. Το απέδειξε στην περίπτωση της Παλαιστίνης τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το λεγόμενο state building. Αν και στην αραβική διένεξη και πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εκφέρει δυνατό πολιτικό λόγο, εν τα τελευταία δύο-τρία χρόνια συμπαραστέκεται στην κυβέρνηση του Προέδρου Αμπάς και του Πρωθυπουργού Φαγιάτ κατά τρόπο που να έχουν οικοδομηθεί οι απαραίτητοι θεσμοί έτσι που μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο ο Πρωθυπουργό Φαγιάτ να είναι σε θέση να ζητήσει από τον οηε την αναγνώριση του ανεξάρτητου κράτους της παλαιστίνης και προσδοκώ ότι όταν αυτή η έκκληση γίνει η ευρωπαϊκή ένωση θα ανταποκριθεί θετικά. η ευρωπαϊκή ένωση θα μπορούσε να διαδραματίσει ανάλογο ρόλο με τις χώρες της περιοχής. εύχομαι και ελπίζω και καλώ την ευρωπαϊκή ένωση να διαπραγματευτεί και να συνάψει σχετικές συμφωνίες με κάθε μια από τις χώρες των οποίων οι λαοί ζητούν αλλαγή και μαζί με τους εκπροσώπους των λαών αυτών να καθορίσουν τους τομείς όπου η ευρωπαϊκή ένωση θα μπορούσε να βοηθήσει οικονομικά αλλά και άλλως πως με την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και τον καθορισμό κοινών προγραμμάτων για την κοινωνικο οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. με τον τρόπο αυτό η ευρωπαϊκή ένωση απαντά και στους στόχους που η ίδια έθεσε στη δική της πολιτική γειτονίας. ευχαριστώ. Ο κ. ο επόμενος, ο για την ελευθερία και δημοκρατία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπατε εκπρόσωπε. Θα ήθελα να επανέλθω σε δύο σημεία το οποίο είπατε ε, και συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε όσον αφορά τι κατευθείαν διαπραγματεύσει, γιατί την περασμένη εβδομάδα είχα την τύχη να κάνω κάποιε μακρέ ε, συνομιλίες με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνηση αλλά και της ΚΝΕΣΕΤ. Βεβαίως θα πρέπει κανείς να δείχνει εμπιστοσύνη στους συνομιλητές του. Αυτοί μιλούν για άμεσες διαπραγματεύσεις με την Παλαιστινιακή Αρχή. Να εξασφαλίσουμε το ότι πραγματικά θα λάβουν χώρα αυτές τις διαπραγματεύσεις. Είναι πολύ σημαντικό για την ειρήνευση. Να εξασφαλίσουμε ότι και οι δύο πλευρές εκπροσωπούνται, κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι. Τώρα έρθει η ώρα να βρούμε αυτό το οποίο θέλουμε, δηλαδή μια αξιόπιστη κυβέρνηση. Να γίνει το μεγαλύτερο προς τα εμπρός. Επίσης, αναφερθήκατε στην μοίρα του επιπενταετή εφραγισμένου Γκίλα Τσαλή και ήρθα σε επαφή πριν λίγες μέρες με τον πατέρα του. Δεν ξέρει Αναρωτιέται. Θα συνεχίσει να πιέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε την απελευθέρωση το σύντομο Το δυνατόν. Ο πρόεδρο. Ε, Φάντερ Στούπ θα ήταν ο επόμενο ομιλητή, αλλά δεν τον βλέπω. Άρα πάμε στον κύριο Πέτερινγκ. Έχετε το λόγο. Κυρία Ήπατη, εκπρόσωπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο αραβικός κόσμος ε, βρίσκεται σε μια ουσιαστική αλλαγή. Οι άνθρωποι αγωνίζονται για την αξιοπρέπειά τους, επιθυμούν να ζήσουν με ελευθερία, δημοκρατία και ευνομία, ακριβώς όπως και εμείς. Είναι λοιπόν ε, πολιτική και ηθική επιταγή για μας ε, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους στον αραβικό κόσμο. Το προηγούμενο Σαββατοκυριακό επισκέφτηκα το Κάιρο και πήγα στην πλατεία Ταχρήρ και συναντήθηκα με πολλούς νέους. Είδα λοιπόν ότι αντιμετωπίζουν το μέλλον με ανοιχτό πνεύμα, με αισιοδοξία και όλα αυτά με επηρέασαν ε, και με εντυπωσίασαν βαθιά. Η Αίγυπτος ε, ε, και άλλες χώρες του αραβικού κόσμου έχουν πλέον την ευκαιρία για δημοκρατικές εξελίξεις. Αυτό αφορά και το Ισραήλ, έτσι ώστε να μην είναι μαζί με το λίγο οι μόνες δημοκρατίες στη Μέση Ανατολή. Η βαθιά αυτή αλλαγή στις αραβικές χώρες είναι μια ευκαιρία για τη διευθέτηση της διένεξης ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Οτιδήποτε παρεμποδίζει την ενευτική διαδικασία πρέπει να ανασταλεί λέει ε, οι επικισμοί είναι πρόκληση για τους Παλαιστίνιους και η πύραυλη της ε, Χαμάς είναι πρόκληση για το Ισραήλ. Πρέπει να σταματήσουν όλα αυτά. Είναι δυνατόν να επιτευχθεί ειρήνη ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Δύο κράτη με ασφαλή σύνορα, καλοί γείτονε που ζουν ειρηνικά. Τώρα λοιπόν δεν είναι η στιγμή για μικροπρέπειες ε, και επιφυλάξεις. Τώρα έχει έρθει η στιγμή για ε, θαραλέες πράξεις. Έχει έρθει η στιγμή για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, για δημοκρατία στις αραβικές χώρες. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ήρθε η στιγμή να δώσουμε και το λόγο στον κύριο Σβόμποντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ας είμαστε λοιπόν ειλικρινείς. Ο μη πόλεμος, γιατί στη Μέση Ανατολή δεν μπορούμε να μιλάμε για ειρήνη, ο μη πόλεμος βασίστηκε στο ότι οι δικτάτορες και τα αυταρχικά καθεστώτα κρατούσαν τους ανθρώπους τους ε, μέσα σε φράχτη αν θέλετε και ε, το ίδιο ίσχυσε και για το Ισραήλ. Βλέπουμε λοιπόν ότι τέτοιου είδους στηρίγματα είναι σαν πύλνα πόδια και καταραίουν. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν ανακατεύτηκε το Ισραήλ στις αραβικές εξελίξεις. Όμως η μία ανάμειξη δεν αρκεί. Όπως είπε ο κύριος Πέτερινγκ, πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία. Το Ισραήλ τώρα πρέπει να δράξει την ευκαιρία να ε, επιτύχει τη μόνιμη ειρήνη που δεν θα βασίζεται σε κάποιους δικτάτορες αλλά σε πραγματική βούληση των λαών να συνάψει ειρήνη. Γι' αυτό λοιπόν οι επικισμοί δεν είναι μόνο αγκάθι, αλλά είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό. Ε, κυρίως ο Υπουργός Εξωτερικών είπε στις Βρυξέλλες ότι μα δεν αφαιρούμε έδαφος ε, από τους Παλαιστίνους Αυτό είναι και διαιρετικό, διχαστικό μάλλον, αλλά και κοινικό. Πρέπει να πάψουν πλέον οι επικισμοί, να ανασταλούν και λυπάμαι που κατέθεσαν βέτο οι Αμερικανοί, γιατί με τον τρόπο αυτό απέδειξαν ότι δεν ενδιαφέρονται πραγματικά, πραγματικά για την ειρηνευτική διαδικασία. Και όταν έγινε λόγος για τις εκλογές, ε, θέλω να αναγνωρίζουμε τις εκλογές ε, ως δημοκρατικό βήμα όχι δηλαδή ε, να αναγνωρίζουμε τους πολιτικούς που βγαίνουν από εκλογές, αλλά μην επαναλάβουμε το λάθος, να αποφασίζουμε εμείς ε, ποια είναι καλή εκλογική νίκη και ποια κακή. Να αναγνωρίζουμε τις δημοκρατικές εξελίξεις και κάτι άλλο, επί το οποίο νομίζω συμφωνούμε όλοι μας. Ελπίζω ότι θα ενισχύσετε τις προσπάθειές σας να μπορεί να επανέλθει ο κύριος Τζαλίτ, επιτέλους να επιληθεί αυτό το πρόβλημα, ε, γιατί όπως είναι κόλλημα η επικιστική σε δραστηριότητες. Το ίδιο ισχύει και η σύλληψη του Τζαλίτ. Νομίζω λοιπόν ότι και τα δύο προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε επιτέλους στη Μέση Ανατολή να έχουμε επικοδομητικές συζητήσεις ε, για την ειρήνη. Ο κύριος Λάμπστορφ, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αντίθεση είναι εντυπωσιακή. Οι αλλαγές στον αραβικό κόσμο εντυπωσιάζουν όλους μας. Ε, προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Συζητήσαμε σήμερα για τη Λιβύη. Τις προηγούμενες εβδομάδες μιλήσαμε για την, την Ισία και την Αίγυπτο. Αλλά τον να υπάρχει παράλληλα ε, αδιέξοδο στην ειρηνευτική διαδικασία και πρέπει να πω κυρία Άστον ότι πραγματικά ήταν επίτευγμα εκ μέρου σας το να επιτύχετε αυτή την τετραμερή. Τετραμερή, ε, έχοντας κατά νου την ανασφάλεια στην περιοχή και στο Ισραήλ. Αυτό πραγματικά ήταν μεγάλη επιτυχία. σα το αναγνωρίζω. Επειδή λοιπόν ακούτε εδώ πολύ συχνά κριτική, καλό είναι να ακούτε καμιά φορά επένου. Όσον αφορά το περιεχόμενο, θέλω να πω με απόλυτη σαφήνεια. Κατά την άποψή μου, το Ισραήλ δεν είναι επιφυλακτικό απέναντι στη δημοκρατία στον αραβικό κόσμο, που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι αλλαγέ. Και εδώ συμφωνώ με τον κύριο Πέτρον και με τον κύριο Σβόμποντα, όταν θα προχωρήσει η δημοκρατία Δημοκρατία, επιτέλου τότε θα υπάρχει και μια μοναδική ευκαιρία να προχωρήσει και η ειρήνη. Πρέπει να ανασταλούν επικιστικέ δραστηριότητε, από αυτού συμφωνούν όλε οι πολιτικέ ομάδε ε, και επίση ε, συμφωνούμε ε, και με τι προσπάθειε συγκάλυψη των γεγονότων. Πάντω, α μην ξεχνάμε το τι συμβαίνει και ε, με τη Χαμάς. Η κατάσταση και στα Παλαιστινιακά εδάφη δεν είναι απλή και εκεί πρέπει να υπάρξει εκδημοκρατισμός. Ε, στην δυτική, ε, στην δυτική όχθη στη Γάζα υπάρχει, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, όμως δεν υπάρχει μετριοπαθής κυβέρνηση και αυτοσυγκράτηση. Η κυρία Νίλσεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Στόρνε, παρατηρώ μια πολύ περίεργη τάση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά τι δηλώσει που κάνουμε για να κατακρίνουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πλευράς του Ισραήλ, εργάζεται το Συμβούλιο για να, εντατικά για να ενισχύσει τις οικονομικές σχέσεις με το Ισραήλ, χωρί να θέτει όρους στι 22 Φεβρουαρίου. De facto αναβαθμίστηκε η Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ και υπάρχουν διάφορες επωνομαζόμενες τεχνικές συμφωνίες για τον ανταγωνισμό, για τις κρατικές προμήθειες, για την ένταξη του Ισραήλ στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και στη Europol, στη Διαστημική Υπηρεσία της Ένωσης κτλ. κτλ. Ε, τέλη Ιανουαρίου ε, ενέκρινε η Επιτροπή τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Ισραήλ, για το οποίο υπάρχουν έχουν υπόνοιες ότι χρησιμοποίησε ευρωπαϊκά διαβατήρια για να διαπράξει μια πολιτική δολοφονία στο Ντουμπάι πέρσι. Ε, πάνω από 800 προγράμματα υπάρχουν ανάμεσα σε πανεπιστήμια και ευρωπαϊκές εταιρείες. Πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις θα δοθούν το 2013 και μεταξύ των δικαιούχων είναι ε, ε, οι κατασκευαστές οπλικών συστημάτων που φτιάχνουν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται κατά της λωρίδας της Γάζας. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτησε τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο κύριος Νετανιάχου για τη Δυτική Όχθη, τη Λωρίδα της Γάζας. Ε, κυρία μου, θα μπορούσατε να μας πείτε για ποια μέτρα διευκόλυνσης μιλάμε, ενώ ε, εκατοντάδες οδηγοί φορτηγών διαδηλώνουν τώρα για να καταγγείλουν το κλείσιμο του περάσματος Καρνή και τι προτείνει ο κύριος Νετανιάχου για να σταματήσει τον επικισμό της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, που προχωράμε εκρηκτικού ρυθμούς. Ε, Τελειώνω, Πρόεδρε. Θέλω να περάσω ένα μήνυμα ελπίδας προ ε, τι εκατοντάδε ε, γυναικών που διαδήλωσαν εχθέ στην Παλαιστίνη. Σας ευχαριστούμε κύριο Λεαρίκα. Ευχαριστώ πρόεδρε κυρία Άστον. Οι αραβικές επαναστάσεις ε, νομίζω συνάδουν με τις ε, φιλοδοξίες των Παλαιστινίων. Αλλά η διαφορά είναι ότι δεν καταπολεμούν τους ηγέτες τους οι Παλαιστινοί. Καταπολεμούν μια κατοχική δύναμη, ξένη δύναμη που τους βάζει φυλακή, τους κλέβει τη γη, τα σπίτια τους, τους βάζει φυλακή, ε, επιβάλλει εμπάργο στη λωρίδα της Γάζας και ένα εκατομμύριο μένουν στους καταβλισμούς προσφύγων παρεμβιάζοντα σε καταφανώ ε, το διεθνέ δίκαιο. Άκουσα τι διευκρινήσει σα, ε, κυρία Άστον, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πιο αυστηρή και πιο κυρίω πιο δραστήρια. Οι αραβικοί λαοί περιμένουν κάτι από εμά. Όλα αλλάζουν τώρα στη Μέση Ανατολή και άρα όλα πρέπει να αλλάξουν ε, και στι κυβερνητικέ αρχέ του Ισραήλ. Θα πρέπει το Ισραήλ να εφαρμόσει το διεθνέ δίκαιο όπω και όλοι οι υπόλοιποι. Χρησιμοποιήστε όλα τα μέσα που έχετε την αμφισβήτηση των συμφωνιών σύνδεση μεταξύ άλλων. Εντάξει για το Σαΐντ, σα σας ρώτησα ήδη τι υποτίθεται να κάνετε για να απελευθερώσετε τον Σαλά Αρμουή, ένα νέο Παλαιστίνιο ε, που σαπίζει στις φυλακές του Ισραήλ εδώ και χρόνια. Ε, επιτέλους, ε, κάντε μια ισχυρή πολιτική δράση, ένα ισχυρό πολιτικό βήμα ούτω ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση αμελητή να αναγνωρίσει το κράτος του Παλαιστινίου με τα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ευχαριστώ. Our Επόμενος ομιλητής ο κύριος Προβέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο βασικός χρηματοδότης της Παλαιστινιακής Αρχής με περίπου ένα δις ευρώ το χρόνο. Ε, και παρόλα αυτά ο πολιτικός ρόλος της Ευρώπης στην ενευτική διαδικασία παραμένει περιθωριακός. Αυτή λοιπόν η μεγάλη οικονομική συνδρομή μας δίνει ε, τη δυνατότητα να ε, ζητάμε στους άμεσα εμπλεκόμενους να επανέλθουν στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Όσον αφορά το θέμα της Παλαιστίνης πρέπει να είμαστε σαφείς. Η ειρηνική συμβίωση με το Ισραήλ δεν θα γίνει μονόπλευρα ε, με το κράτος της Παλαιστίνης ε, που μεταξύ ούτε καν και αυτό δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Πρέπει ε, να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, να λυθούν τα προβλήματα κυρίως όσον αφορά τα ασφαλή σύνορα, το, την πόλη του, της Ιερουσαλήμ και το καθεστώς των προσφύγων. Ακόμα και μια μερική συμφωνία θα ενίσχυε τη θέση και των δύο πλευρών και θα περιόριζε τις ακραίες πράξεις, ε, τους εξτρεμιστές. Η κυρία Ντότζ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε κυρία Υπάτη Εγώσοβη. Τα σήματα των καιρών, το σημείο των καιρών είναι ο εκδημοκρατισμός και κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί στους λαούς της Νησίας, της Αιγύπτου και τώρα της ε, Λιβύης το, αυτό που αξίζουν δηλαδή ελευθερία και δημοκρατία. Συμφωνώ με την υπάτη εκπρόσωπο ότι αυτά τα γεγονότα δεν αποστρέφουν την προσοχή, αντίθετα μας επιβάλλουν, τον εστιάζουμε ε, με καινούριο βλέμμα, καινούριο φρέσκο μάτι την προσοχή μας που γίνονται εκεί. Γιατί στο παρελθόν είχαμε την εμπειρία το τι έγινε όταν υπήρξε πολιτικό κενό. Ήρθε η Χαμάς και η Χεσμπολάχ. Άρα θα πρέπει να κάτσουμε και να δούμε πώς μπορούμε τον καλύτερο τρόπο να βοηθήσουμε και για την ειρηνευτική διαδικασία και για την σταθερότητα θα πρέπει να αναγνωριστεί το ότι πραγματικά χρειάζεται ασφάλεια, χρειάζεται κάποιες συμφωνίες ε, σωστές με τις γειτονικές χώρες και να προσέξουμε πού δεν πετύχαμε στην ε, ε, πολιτική γειτονία. Μετά από 1,5 δις το οποίο έχουμε διασπαθήσει για την πολιτική γειτονία, ε, ας κάτσουμε τώρα για να δούμε, κερδίσαμε τίποτα. Έχουμε δεκάδες χιλιάδων που συνέχεια ε, προστίθεται στην αγορά εργασία, δεν έχουν ε, στην Αίγυπτο μέλλον. Θα πρέπει άρα να κάτσουμε και να σκεφτούμε ότι εν σπέρματι μια καινούργια επανάσταση εν υπάρχει. Μιγιάν Μον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Σεπτέμβριο του 2011 θα θέλαμε πραγματικά να ολοκληρωθούν οι ε, επαφές και να πάμε σε μια ειρήνη. Όμως ε, οι προοπτικές δεν δείχνουν να ευωδώνεται αυτή η ευχή γιατί έχουμε τα θέματα των επικισμών. Νομίζω ότι αν χάνεται χρόνος ούτε ο σκοπός επιτυγχάνεται ούτε ε, συμφέρει και το Ισραήλ. Άρα θα πρέπει να βρούμε κάποιους μετριοπαθείς ηγέτες στην Παλαιστίνη που να έχουν την υποστήριξη και την νομιμοποίηση για να κλείσουν συμφωνία με το Ισραήλ. Και αν ε, συνεχιστούν έτσι οι επικισμοί πάρα πολύ δύσκολα θα έχουμε βιώσιμο παρεσθενικό κράτος. Συμφωνώ με σας κυρία Υπάτη ε, δεν θα πρέπει να επηρεαστεί η διαδικασία της ερήνευσης από την αναστάτωση στην περιοχή. Ε, θα πρέπει να έχουμε σε αυτές τις χώρες τώρα δημοκρατικές κυβερνήσεις, οπότε ε, τελικά θα υπάρξει πίεση και για το Ισραήλ. Ίσως θα απομονωθεί ακόμη περισσότερο από τις ε, γειτονικές αραβικές χώρες. Όλοι και το Ισραήλ θέλουν το συντομότερο επομένως. Συμφέρει το συντομότερο μια λύση. Το συντομότερο. Και έτσι να πάμε προς την ολοκλήρωση της ειρήνευσης. Σε συνεργασία και με το Κορτέτο και με τις είπα Συνεχίστε επομένως όπως ε, είχατε πει στο μόναχο με τη δήλωσή σας. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ντερόσο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση στην περιοχή εγκυμονεί κινδύνους ε, και ελπίδες. Ε, οι δημοκρατικές ε, κινήσεις γύρω από το Ισραήλ βεβαίως είναι ευκταίες, αλλά πρέπει να αποφύγουμε τα στραπ που τις αντιμετωπίζουν ως απειλή. Πήγα στη Γάζα το Δεκέμβρη και η πιο συγκινητική ιστορία ήταν του μικρού παιδιού που πήγαινε τα παιχνίδια του κάθε μέρα στο σχολείο γιατί δεν ήταν σίγουρο κατά πόσο θα γύριζε πίσω το βράδυ στο σπίτι του, θα έβλεπε τους γονείς του και το σπίτι του. Αυτό το παιδί λοιπόν θέλει την ειρήνη. Όλοι επιθυμούν στην περιοχή να έχουν ασφαλή σύνορα του Ισραήλ ε, και της Παλαιστίνης με βάση τη γραμμή του 57. Επίσης ε, πρέπει να σταματήσουν οι επικισμοί. Είναι απαράδεκτο ότι ο κύριος Νετανιάχου απορρίπτει τις εκκλήσεις από όλου του του Ισραήλ να αναστείλει τους επικισμούς. Όχι να τους ε, κατεδαφίσει, να τους αναστείλει αυτό είναι απολύτω απαραίτητο για να ξεκινήσουν σοβαρέ διαπραγματεύσει. Είναι προπόθεση και απευθύνομαι έκκληση στην κυρία Άστον ε, να μεταβιβάσει και αυτή περαιτέρω την έκκληση αυτή στου Ισραηλινού. Παρακαλώ, αναστείλετε του επικισμού για να ξεκινήσουν οι συζητήσει ο ε, Πρωθυπουργός Φαγιάντ ε, μπορούν να οδηγήσουν ειρηνικά τους Παλαιστινίους σε Παλαιστινιακό κράτος. Δεν γνωρίζουμε ε, ποιες θα είναι οι συνέπειες αν δεν γίνει κάτι τέτοιο σύντομα. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Ντέιβις δεν μπορούν να είναι μεγαλύτεροι φίλοι του Ισραήλ ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τους Γερμανούς. Η κυρία Μέρκελ λέει στον κύριο Νιτανιάχο εσείς δεν κάνατε τίποτα για να προωθήσετε την Ελληνική. Δώστε μου κάτι, κάτι να έχω κι εγώ στα χέρια μου. Και έχει βεβαίω δίκιο. Το Ισραήλ ε, θέλει να κερδίσει χρόνο. Χρόνο κάνει συζητήσεις για τις συζητήσεις γιατί αυτός ο χρόνος του δίνει τον, τη δυνατότητα να αλλάξει ε, πράγματα επίτόπου επί της ουσίας. Ε, κυρία, είπα ύπατη έχετε την εξουσία να επιφέρετε αλλαγέ. Υπήρξε μία δήλωση πριν από λίγο καιρό, έξι σελίδες καταδίκης ε, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, παραβιάσεων από πλευρά του Ισραήλ και παρόλα αυτά στο τέλος που καταλήγεται λέγεται θέλουμε την καλύτερη και στενότερη συνεργασία με το Ισραήλ. Μα τι κάνετε εδώ, τι είναι αυτό. Ε, είναι σαν να έχετε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Κυρία Ήπατη εκπρόσωπε, εσείς ε, μοιάζει να έχετε έναν ευχάριστο διάλογο, αλλά το Ισραήλ πιστεύει ότι είμαστε αδύναμοι. Αν λοιπόν δεν χρησιμοποιήσετε την εξουσία σας, τίποτα δεν θα αλλάξει. Και γι' αυτό εκείνη τη λέξη που πρέπει να χρησιμοποιήσετε απέναντι στο Ισραήλ είναι ένα όχι, ένα ηχηρό όχι. Κύριο κύριος Κάμπελ Μπάνερμαν, τώρα πάλι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, βομβαρδίζεται, βομβαρδίζεται ο λαός του, της Λιβύης από τον κύριο Καντάφη και ταυτόχρονα βλέπουμε κάποια σχέδια της ε, Λιβύης να ενισχύσει την τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Ε, προτίθεται ο κύριος Καντάφη. Καταλαβαίνετε και ζητούνται επιπρόσθετα, επιπρόσθετη πέρα από τα τρία δις που αναμένεται να αναλάβει η υπηρεσία εξωτερική ε, ε, δηλαδή βλέπουμε ότι αυτή η υπηρεσία ε, εξωτερικής δράσης ρουφάει διαρκώς κονδύλια, 48 εκατομμύρια λίρες τερλίνες πληρώνουμε εμείς για να υπερασπιστεί η Ένωση τα δικά της τα συμφέροντα και θέλουμε να έχουμε σε εμπόλεμες ζώνες αεροπλανοφόρα και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Ε, ε, ζητώ ε, τουλάχιστον ε, θυμηθείτε τι έχει γίνει την εποχή της κυρίας Θάτσερ. Δεν πρέπει να υποπέσουμε στα ίδια λάθη. Ο κύριος Πρέντα, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ε, μιλήσω για τους απεσιόδοξους, ε, για τους σκεπτικιστές ε, που ισχυρίζονται ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη λεκάνη της Μεσογείου η παράπλευρη απώλεια θα είναι η ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής. Η ειρηνευτική διαδικασία ενδέχεται να εκτροχιαστεί ενώ ήδη έχει καταλήξει τώρα σε ένα τέλμα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είμαστε τόσο απεσιόδοξοι γεγονότα, τα πρόσφατα γεγονότα δείχνουν ότι θα πρέπει να επενδύσουμε στην ειρηνευτική διαδικασία και ε, χρειάζεται ο ηγετικό ρόλο Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε ε, να τηρηθεί η καταλεκτική προθεσμία, δηλαδή ο Δεκέμβρη του 2011. Ευχαριστώ την ύπατη εκπρόσωπο για την αφοσίωση που δείχνει και για τι προσπάθειε που έκανε του τελευταίου μήνε, ούτω ώστε να επιτύχει αυτή τη λύση των ε, δύο κρατών και για να έχει μια συνολικότερη ειρήνη στην περιοχή. Χρειαζόμαστε και τι δύο πλευρές τραπέζι των διαπραγματεύσεων και η πρωτοβουλία του να διαβουλευόμαστε χωριστά με τους ε, Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους διαπραγματευτές είναι μόνο ένα πρώτο βήμα, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Οι εξελίξεις στη Μεσόγειο ενδέχεται και να τονώσουν την ε, ειρηνευτική διαδικασία, αλλά οι αλλαγές δεν θα πρέπει να οδηγήσουν ε, σε αναθεώρηση παλιών συμφωνιών με το Ισραήλ. Πρέπει να προσέξουμε. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Σασόλη τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι. Η Μεσόγειος ε, έχει μπει με, με, με δύναμη, με φόρα στην μέση διάταξη της πολιτικής μας. Ε, δεν επενδύσαμε σε πολιτική για τις χώρες Μαγκρέμπ. Εμεί ε, δεν θελήσαμε να εφαρμόσουμε μια κοινή πολιτική για τη μετανάστευση. Αυτό που συμβαίνει στην Βόρεια Αφρική οδηγεί στο να συμπεράνουμε ότι η ειρηνευτική διαδικασία αναγκαστικά θα πρέπει να αναστελεί. Όμω θα πρέπει να βοηθήσουμε του Ισραηλινούς και του Παλαιστίνιου να συμμετάσχουν στι διαπραγματεύσει. και αυτό με βάση προτάσει ε, από κοινού από το Συμβούλιο ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, πολλοί κάνουν έκκληση στο Ισραήλ να αλλάξει στάση, να συνδυάσει την ασφάλεια με την ειρήνη. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να σκίσει πίεση στο Ισραήλ για να χαλαρώσει την πίεση στα κατεχόμενα, να αναστείλει την την πολιτική των επικισμών. Αυτός απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Ε, όταν ε, πνέει ε, άνεμος ελευθερίας, όλοι καταλαβαίνουμε ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση οδηγεί σε κίνδυνο το να μην λάβουν σάρκα και οστά οι ελπίδες των πολιτών θέτουν όλα αυτά σε κίνδυνο τις προοπτικές ε, τόσο για τη Μεσόγειο όσο και για τη Μέση Ανατολή προοπτικές που είναι πάρα πολύ ευαίσθητες. Όλοι βλέπουμε πώ αλλάζουν τα πράγματα στην ε, Αγγλική Ανατολή ε, και πώ η δημοκρατία διαδικασία, Μαγκρέπ, Μασουράκ, Αίγυπτο κατησχύουν και επομένω βλέπουμε τι έγινε σε σχέση με το Ισραήλ και με τους Παλαιστίνιους θα πρέπει να το δουν έως όχι σαρίς σαν ευτυχία και εγώ πιστεύω ότι αυτή η δημοκρατική εξέλιξη για τους Παλαιστινίους είναι μια ευκαιρία που θα πρέπει και οι μεν και οι δε να την αρπάξουν διότι σήμερα και οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνοι έχουν μπροστά τους μια πραγματικότητα ε, αλλάζει ο κόσμος γύρω τους ήρθε η ώρα επομένως και αυτοί να κινηθούν ε, και επομένως ε, και η Ευρώπη θα πρέπει να του εξωθήσει προ διάλογο αυθεντικέ διαπραγματεύσει και να αρχίσει μια πραγματική διαδικασία ειρήνευση που θα καταλήξει σε μια βιώσιμη λύση για αυτά τα, τα, τα κράτη που θα πρέπει να συνεπάρξουν ειρηνικά. Όμω σε μια τέτοια κρίσιμη συγκυρία ε, είναι άστοχο ε, το να μην υπάρξει ε, ειδικό απεσταλμένο. Οπότε θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε το, το τι θα γίνει όσον αφορά αυτό. Και σα ευχαριστώ και τον πατέρα. Εμεί ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρο. Και τώρα δίνει τον λόγο στον κύριο Λίσεκ. Κυρία Υπάτη εκπρόσωπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ήδη μου έχει δοθεί ευκαιρία τους τελευταίους μήνες να επισκεφθώ μια σειρά χωρών της Μέσης Ανατολής, της Αγγής Ανατολής, ε, Συρία, στην Παλαιστίνη, στο Ισραήλ και ε, κάποιος από τους ε, ηγέτες μου είπε ότι θα πρέπει η Ευρώπη να ασχοληθεί περισσότερο. Πρόκειται για μια επένδυση που αν ε, αποδώσει θα είναι μια επιτυχία μεγέθους άξια για ένα νόμπελ. Αυτό θα μας πω κύριε Πρόεδρε. Όμως ε, όλοι λένε το ίδιο. Όλοι οι άνθρωποι από εκεί λένε το ίδιο. Περισσότερο να ασχοληθεί η Ευρώπη στην ε, Μέση Ανατολή υπάρχουν ε, προβλήματα, δεν μπορεί να ασχοληθεί περισσότερο η Αμερική. Όμως θα πρέπει εμεί να ασχοληθούμε περισσότερο, θα πρέπει να συνεργαστούμε και με τις ΕΠΑ. Ε, είναι στατική σημασία ε, η υπόθεση αυτή, οπότε θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία που δίνετε τώρα. Γιατί ξέρετε την περασμένη εβδομάδα μόλις είχαμε συνάντηση μεταξύ Ισραηλινών και πολωνικής κυβερνήσεως. Σε επίπεδο πρωθυπουργών πήγε στο Ισραήλ ο κύριο Σικόρσκι. Αυτό δεν είχε προηγούμενο. Θα πρέπει με αυτήν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε. Πάσκο. Το θέμα της ε, Μέσης Ανατολής είναι περίπλοκο, αλλά έχει περιπλακεί περισσότερο τώρα τελευταία. Το καλύτερο για όλους ήταν να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ε, ε το θέμα είναι για τους ε, Παλαιστίνιους ποιος θα τους βοηθήσει. Η Χαμάς επεκτείνεται περισσότερο. Ε, είναι πιθανόν η Φατάχα να κερδίσει το πάνω χέρι. Αυτό δεν μοιάζει πιθανόν. Ε, η Ορδανία και αυτή μπορεί να ανατινάξει την ειρηνευτική διαδικασία. Για το Ισραήλ υπάρχουν δύο σχολέ σκέψη. Η μία είναι υπέρ τη επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μέσα από ρηξικέλευτε προτάσει και άλλοι πάλι λένε ότι πρέπει να συνεχιστεί η ίδια πολιτική. Πάντω με όραμα και αποφασιστικότητα μπορούμε να βοηθήσουμε να υπάρξουν εξελίξει ε, και μπορεί να ξεπεραστεί το αδιέξοδο που υπάρχει αυτή τη στιγμή ή βεβαίως ε, μπορεί τελικά να αποδειχθούν και όλα αυτά ε, αυταπάτη. Και τώρα το λόγο έχει η βεβαιως μπορει τελικα να αποδειχθουν και ολα αυτα αυτα πατη και τωρα το λογο εχει η κυρια γιαννακου για 1,5 λεπτό. Ε, συμφωνώ με τις, τα σχόλια της υπάτης εκπροσώπου ότι τώρα είναι η στιγμή για να υπάρξει ουσιαστικότερη παρέμβαση ε, για μια σωστή διαπραγμάτευση στη Μέση Ανατολή ε, πρώτον γιατί δεν γνωρίζει κανείς την εξέλιξη που θα υπάρξει στις χώρες της βορείου αφρικής και δεύτερον διότι είναι σαφές ότι η κατάσταση ανάμεσα στο ισραήλ και την παλαιστίνη είναι αυτή που χρησιμοποιείται ως άλοθη και για την τρομοκρατία και για εντάσεις σε όλο τον κόσμο και για πυροδότηση ειδικότερα εντάσεων στο μουσουλμανικό κόσμο. επομένως η ειρηνευτική διαδικασία χρειάζεται άμεση παρέμβαση δική σας κυρία ε, εκπρόσωπε και ειδικού απεσταλμένου και θα είναι και μια άσκηση για την ευρώπη για να δούμε αν πραγματικά μπορεί να παρέμβει και να παίξει το ρόλο που έπαιζαν οι ηνωμένε πολιτείε με άλλοτε άλλα αποτελέσματα. φυσικά η οικονομική βοήθεια είναι απαραίτητη αλλά χρειάζεται ειδική ρύθμιση και ειδική παρακολούθηση γιατί είναι γνωστό τι είχε γίνει με την οικονομική βοήθεια σε προηγούμενες εποχές. και βέβαια είναι το τεράστιο θέμα τη δημοκρατική συγκρότηση γιατί χωρίς δημοκρατική και κοινωνική συγκρότηση ασφαλώς και η ειρηνευτική διαδικασία καθίσταται πολύ δύσκολη. έτσι ένας ειδικός διαπραγματευτής με μια ειδική ομάδα η οποία θα είχε σχέση και με τη δημιουργία μιας ουσιαστικής δημοκρατικής συγκρότησης και συνταγματικής τάξης θα είχε ιδιαίτερη αξία κυρία εκπρόσωπε και έχω την εντύπωση ότι αυτή την προσπάθεια με βάση αυτά που είπατε θα την αναλάβετε. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα θα μιλήσουμε με την Κυρία Κολάρσκα-Μπομπίν. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συναδελφοί. Για τις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής ακούμε συχνά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι παίκτη σε αυτή τη σκηνή. Ε, είναι αυτός που πληρώνει και μόνο. Ε, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει και τους δύο ρόλους. Ε, θα πρέπει να διαδραματίζει το ρόλο της όχι μόνο να ε, εκταμιεύει κονδύλια. Η Επίσης ε, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η θέση της ε, Ρωσίας. Ε, κάποιοι περιμένουν μια θετική δράση από τις ΗΠΑ Ε, και για την ε, ε, επίλυση, τη λήξη της σύραξης οφείλουμε να δράξουμε αυτή την ιστορική ευκαιρία που έχουμε τώρα. Διαθέτουμε εδώ και την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ανοιχτή μη το εργαλείο και μπορούμε να έχουμε μια κοινή πολιτική στον τομέα αυτό. Δημοσιεύθηκε ένα έγγραφο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά ε, με ε, την ε, μεσογειακή συνεργασία, τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις μεσογειακές χώρες, νομίζω ότι θα πρέπει η στάση μας στην Μέση Ανατολή να συνάδει με την πολιτική που ακολουθούμε γενικότερα για τις μεσογειακές χώρες. Υποστηρίζεται με τις δράσεις μας η κοινωνία των πολιτών, η ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής και στο παρελθόν. Έχουμε κάνει τόσα πολλά πράγματα, θα χρησιμοποιήσουμε για να εκπονήσουμε τη μελλοντική μας πολιτική. Κυρία Μουσκουαρντίνη. Κυρία Υπατή εκπρόσωπε, η ειρήνη έχει ανάγκη από δεσμεύσεις τις οποίες πρέπει να λάβουν όλοι. Ξεκινάμε από την αναγνώριση του Ισραήλ, κάτι το οποίο όμως δεν υπάρχει ακόμα, τουλάχιστον όσον αφορά κάποιες χώρες. Και γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο απαραίτητο για να υπάρξει ειρήνη όλες οι χώρες περιοχής να προσφέρουν τις ελάχιστες ε, προϋποθέσεις, τις απαραίτητες, έτσι ώστε οι σχέσεις να βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό. Σήμερα η εμπορική πολιτική είναι μια νέα μορφή εξωτερικής πολιτικής και αυτό ε, δεν αφορά μόνο τη δημοκρατία, αλλά αφορά και τις εμπορικές ε, σχέσεις που και εκεί πρέπει να αναστηθούν κάποιες λύσεις. Δεν είναι πλέον δυνατόν, όπως συνέβη μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να χρηματοδοτεί προγράμματα ε, όπου δεν προκύπτει το αναμενόμενο αποτέλεσμα ούτε προκύπτει έστω και αργή ε, βελτίωση της ε, δημοκρατικής διαδικασίας και της ειρηνευτικής. Το Ισραήλ δεν μπορεί να φεθεί στη μοίρα του ο Παλαιστινιακός λαός, λαός από την πλευρά του έχει δικαίωμα σε κράτος. Ως εκ τούτου εμείς πρέπει να παρέμβουμε σε οικονομικό επίπεδο με παρατηρητές που είναι σε θέση να παρακολουθούν την χρήση των κονδυλίων μας ε, το ότι επενδύουμε σε μια μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή αυτό επιτέλους επιβάλλει στην Ευρώπη να αναλάβει μια πιο ισχυρή και αποφασιστική πρωτοβουλία να συμμετάσχουν περισσότερο και οι νέοι οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν έτσι ώστε να οικοδομηθεί μια πιο ασφαλής και δημοκρατική κοινωνία κάτι το οποίο εμείς δεν μπορέσαμε να προσφέρουμε στις νέες γενναίες. Πολύ ωραία. Λέω, ο Πρόεδρος, τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία Catch the Eye ε, και όπως είχα αποσχεθεί δίνω το λόγο πρώτα απ' όλα στον κύριο Αλάχη. Μία ερώτηση προς την ε, κυρία Άστον άκουσα αυτά που μας είπατε και έχω να σας υποβάλω δύο ερωτήσεις που έχουν σχέση με τη δική σας την αξιολόγηση ε, για την στασιμότητα, το αδιέξοδο στην ειρηνευτική διαδικασία και σε αυτά που συμβαίνουν τώρα στη Βόρεια Αφρική. Δεν πιστεύετε κι εσείς ότι μας προσφέρονται νέες ευκαιρίες ε, ε, τη στιγμή που τώρα ε, οι απαιτήσει ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ πιο ουσιαστικές και είναι σαφέστερα τα κριτήρια για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων όμως βλέπουμε ότι χαμηλώνουν τα κριτήρια, χαμηλώνουν τα κριτήρια για τις παραβιάσεις στη Γάζα παραδείγματος χάρη. Εξάλλου δεν πιστεύετε ότι η πολιτική του Ισραήλ του παρελθόντος τώρα πλέον δεν δικαιολογείται διότι η Κνεσέτ ε, είναι όλο και λιγότερο δημοκρατική και οι δημοκρατίες βασικά δεν μπαίνουν σε πόλεμο. Όλα αυτά εσείς τι θεωρείτε ότι βελτιώνουν στην ύφεση στη Μέση Ανατολή. Βλέπω ότι και ο κύριος Τάνοκ θέλει να λάβει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εγώ ε, ήθελα να μιλήσω για ένα λεπτό στο κάτσου Δεν θέλω να κάνω ερώτηση. Έχω το λεπτό μου. Ωραία. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέρος ε, του, ε, της τετραμερούς, αλλά δεν υπάρχει μεγάλη πρόοδος ε, στη σχέση με τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους. Το αδιέξοδο θα παραμείνει όσο εξακολουθεί να υπάρχει ανασφάλεια στον αραβικό κόσμο. Από το πρίσμα του Ισραήλ και εγώ δηλώνω ότι είμαι αντιπρόεδρος ε, του Ευρωπαϊκού Κύκλου Φίλων του Ισραήλ. Έχουμε μια παράδεκτη κατάσταση. Η Αίγυπτος είναι εκείνη που ε, αποσπά την προσοχή από την ειρηνευτική διαδικασία. Εγώ λοιπόν απευθύνθηκα στην κυβέρνηση και τους είπα να ε, σεβαστούν σεβαστούν τη συμφωνία του 79 με το Ισραήλ ε, και οι αδελφοί μουσουλμάνοι και αυτοί να σεβαστούν αυτή τη συμφωνία. Αυτό που χρωστάμε στην Αίγυπτο είναι ε, ε, να συμβάλλει στην ευτική διαδικασία με το Ισραήλ. Δυστυχώς όμως κυβερνάει η Χαμάς ε, η οποία είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο για την ειρήνη και το Ιράν αποτελεί μια μεγάλη απειλή για το Ισραήλ. Η ειρήνη στην περιοχή δεν θα είναι ποτέ δυνατή όσο η Τεχεράνη συνεχίζει να χρηματοδοτεί τους φανατισκούς της Χεσμολά στο Λίβανο. Γι' αυτό λοιπόν κατανοώ την ανησυχία του Ισραήλ όταν είδε να περνάνε τα σκάφη από τη Συρία η Αίγυπτος πλησιάζει το Ιράν και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Γι' αυτό λοιπόν εύχομαι στην είπατη εκπρόσωπο καλή επιτυχία σε αυτό το διπλωματικό ναρκοπέδιο στο οποίο καλείται να περπατήσει. Ήρθε η σειρά του κυρίου Πάσκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή ε, βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει λοιπόν ε, να ε, προβλέψουμε πώς ακριβώς, ποια θα είναι τα μελλοντικά καθεστώτα και στις δύο αυτές ε, χώρες να εμποδίσουμε τις προσπάθειες του Ισραήλ να οικοδομήσει νέους οικισμούς στα Παλαιστινιακά εδάφη. Είναι μονόδρομος Η μοναδική λύση είναι να συμμετάσχουν και οι δύο πλευρές και να πείσουμε τις δύο πλευρές να απόσχουν από οποιοδήποτε δραστηριότητες εξοργήσουν ε, τους ε, λαούς των αραβικών χωρών. Ε, δεδομένων και των τελευταίων εξελίξεων οφείλουμε να μεριμνήσουμε ώστε να ανέβουν στην εξουσία αξιοπρεπείς δημοκρατικές δυνάμεις ούτως ώστε χωρίς μίσος, χωρίς εμπάθεια να λήξει αυτή η διαμάχη, αυτή η σύρεξη. Πιστεύω ότι κατάλαβε πλέον η Ισραηλινή κυβέρνηση ότι ήρθε η στιγμή να εισέλθει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με τους Παλαιστινίους. Ο κύριο Φόμποντα, τελευταίο ομιλητή. Ο κύριο Τάνοκ είπε ότι τα σκάφη του Ιράν πέρασαν από το Σουέζ και γι' αυτό λοιπόν ερωτώ την κυρία Αστον. Είναι εξασφαλισμένο ότι αυτό έγινε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Δεν υπήρχε πραγματικά καμία δυνατότητα για την Αίγυπτο να απαγορεύσει τη διέλευση αυτή. Είτε δεν ερωτώ αν άρεσε ή όχι στην Αίγυπτο, αλλά ερωτώ κατά πόσον υπάρχει μια πολιτική προέκταση σε αυτό το γεγονός που έλαβε χώρα. Νομίζω ότι η κυρία Άστον ε, κατέγραψε όλες τις που που έτσι και τώρα πλέον έχει το χρόνο για να απαντήσει. Θα προσπαθήσω, Πρόεδρε, να απαντήσω σε όσο γίνεται περισσότερες ε, ερωτήσεις. Αλλά πάντοτε όταν συζητούμε την ενευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, τότε όλοι ε, συναισθανόμαστε το πόσο επίγουν τα πράγματα, το πόσο προσδοκούμε όλη την επίτευξη κάποιας πρόοδου. Και σας διαβεβαιώ ε, ότι κάνω ό,τι μπορώ και προσπαθώ να πετύχουμε κάτι από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι και δεν θέλω να, να, να ακούσω όμως ξανά να μου λέτε ότι εμείς μόνο πληρώνουμε και δεν είμαστε παράγον παίκτη στην περιοχή, στο θέατρο αυτό των εξελίξεων. Δεν θέλω να σας φημώσω, αλλά όχι μην το ξαναλέτε αυτό. Προσπαθούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και επιτόπου και θα σας εξηγήσω. Εγώ θέλω τώρα να αρχίσω με αυτά που είπε ο κύριος Σαλαφράγκα γιατί μου ζήτησε κάποιες συγκεκριμένες διευκρινήσεις όσον αφορά αυτή την άρνηση κυρία του Συμβουλίου Ασφαλείας αυτό το 14-1 με το βέτο τον είπα όσον αφορά τους ε, επικισμούς σε σχέση με το ψήφισμα εκείνο του Λιβάνου που τότε ήταν στο Συμβούλιο Ασφαλείας όμως ε, ε, προκάλεσε πολλούς κλειδονισμούς, πολλές διαταράξεις του ΣΥΠΗΝ και ε, είχαμε αγανάκτηση και όπως ξέρετε όλοι ήταν κατά των Αμερικανών και εμείς το ίδιο τώρα η θέση μας είναι κρυστάλλινη όλοι είμεθα ενωμένοι και αναγνωρίζουμε ότι είναι παράνομη είναι κατά του διεθνούς δικαίου αυτή η επικισμή. Και προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι κανένα δεν συμφέρει να υπάρχουν εκεί πέρα και θα πρέπει τελικά το πρόβλημα αυτό να επιληθεί με καθορισμό των σενόρων. Και είπαμε εμείς για τα σύνορα του 67 να το συμφωνήσουν είπαμε, μεταξύ τους οι εμπλεκόμενοι. Δεν μπορούμε να τους το επιβάλλουμε. Αλλά θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πραγματικότητα που ζει ο καθένας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα για τις μακρόπνες σχέσεις με τις ΕΠΑ και κύριε ξέρετε οι ΕΠΑ έχουν πάρα πολύ σκληρά προσπαθήσει να εξηγήσουν γιατί έκαναν αυτό το οποίο έκαναν και εγώ συνεχίζω να συνομιλώ και με τους Αμερικανούς και με τους Παλαιστινίους οι οποίοι νομίζω ότι έχουν αντιληφθεί γιατί έγινε αυτό που έγινε. Επομένως πάρα πολλά θα πρέπει ακόμα να γίνουν και με τίποτα δεν σας λέω ότι ε, τα πράγματα ήταν εύκολα. Με ρωτήσατε για τις ε, Παλαιστινιακές εκλογές για το Σεπτέμβριο που η Χαμάς αρνείται να συμμετάσχει. Είδατε τι έγινε, είδατε ο κ. Φαγέντ προσπαθεί να δει πώς μπορεί να συμφιλιώσει τα πράγματα. Θα του μιλήσω σύντομα και γι' αυτό αλλά και για πολλά άλλα. Δεν ξέρω τι θα γίνει τόσο πρώτα εκλογές ας Α αποφασίσουν οι Παλαιστίνοι αναζητούν την καλύτερη δυνατή λύση. Επίσης μου είπατε αυτό έχει σχέση με το Wikileaks, τις, τις διαρροές ε, για τους Παλαιστινίους και ξέρω ο κύριος Έρκατ που ήταν ο επικεφαλής της διαπραγματεύσης, τώρα έχει αλλάξει θέση, τώρα έφυγε από εκεί που ήταν ε, και το αποτέλεσμα ήταν πρώτα πρώτα μεγάλος προβληματισμός για το τι γίνεται γιατί όταν προσπαθείς να βρεις μια θέση για προδιαπραγμάτευση πάρα πολλά λέγονται και πολλά από αυτά που λέγονται δεν αποκρισταλώνονται στο τελικό κείμενο και ενδιάμεσα ο κόσμος σκέφτεται και, και προβληματίζεται επομένως πολλά ελέγχθησαν και για τη Δυτική Όχθη και άλλα όμως παρουσιάζει ενδιαφέρον το υπήρχε και αντίθετη αντίδραση νομίζω ότι στο Ισραήλ κάποια ΜΜΕ ε, είπανε Καλά, αφού είναι έτσι εμείς γιατί έχουμε παρασυρθεί. Άρα ήταν περίεργος ο ενδιαφέρον προβληματισμός και ίσως μακροπρόθεσμα, αν και ποτέ δεν είναι υπέρ των ε, διαρροών, γιατί οι σωστές πολιτικές έτσι εμποδίζονται και μακρόπνοα ε, δεν θα αποδώσουν οι καρποί ε, όπως στην αρχή φάνηκε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα όσον αφορά την Συμφωνία Σύνδεσης τι έγινε, μάλλον τι δεν έγινε, δεν έγινε τίποτα, δεν άλλαξε με τίποτα το πλαίσιο. Η πρόοδος συνεχίζεται και θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον η ενευτική διαδικασία επίσης ε, προχωράει. Ελέγχθη ότι θέλαμε να έχουμε στενές σχέσεις και πιστεύουμε ότι θα πάμε για δύο κράτη. Θέλουμε οικονομικά, πολιτικά να ενισχυθούν τα κράτη αυτά και η Παλαιστίνη και το Ισραήλ. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι εμείς θα προχωρήσουμε στην ε, συμφωνία σύνδεσης εάν δεν προχωρήσει η ειρήνευση. Ε, επίσης, ε, πάρα πολύ σωστά λέξη θα πρέπει να επιταχύνουμε τις εξελίξεις για με τους μεν και με τους δε και επίσης να ληφθεί υπόψη το ότι υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην περιοχή όπως και ο υπάρχουν αλλαγές που απαιτούν να αναγνωρίσουμε ότι έχει καινούργιο ρόλο η Αίγυπτος. Όχι, δεν λέω ότι θέλει τώρα σπατιωτικά κάτι να κάνει κατά του Ισραήλ η Αίγυπτος. Καθόλου δεν το πιστεύω αυτό. Αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Αίγυπτος τώρα θα τα πάει καλύτερα και είναι στο, στο, στο, στο περιβόλι τους των εμπλεκομένων. Να, λοιπόν, γιατί όλοι έχουν συμφέρον εξέβρεσης λύση. Έτσι θα αποκτήσει σταθερότητα η περιοχή και ασφάλεια. Το έλεγα και το λέω. Και θα το λέω σε όλους. Και στο κόρτετο. Ναι κύριε Μπέλτερ, όντως θα πρέπει να πάμε εκεί για τις διαπραγματεύσεις, αλλά να είμαστε σίγουροι ότι είναι αξιόπιστοι οι διαπραγματευόμενοι. Α, εκεί είσαστε, συγγνώμη, συγγνώμη, κοίτα γαλλού, αλλάξατε θέση. Επομένως θα πρέπει να πάνε οι Παλαιστίνα κατά των διαπραγματεύσεων και ο Αραβικό Σύνδεσμος να του στηρίξει. Τα είπαμε την Αραβικό Σύνδεσμο στο Κάιρο, 14 Μαΐου. Ε, αυτός ο συνομιλητής μου θα είναι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές στην Αίγυπτο. Όμως είναι σημαντικό να υπάρχει λαϊκή νοημοποίηση για τις διαμετεύσεις των Παλαιστινίων. Όλα αυτά επομένω ε, αλληλεξαρτώνται και άρα θα πρέπει να διαμορφωθεί μία πεποίθηση για το κατά πόσον αυτό θα σχέσει για όλους. Κύριε Λάμπστοφ, ευχαριστώ για όσα είπατε. Ναι, το κορτέτο είναι κάτι πολύ σημαντικό σαν φορέας ας πούμε, αλλά δεν είναι πανάκια. Και εγώ πιστεύω 100% ότι έχουμε διδαρματίσει σημαντικό ρόλο. Και συνεχίζουμε να παίζουμε σημαντικό ρόλο τελευταίους μήνες και εβδομάδες. Και έτσι τα πράγματα να μην αποτελματώνονται. Όμως θα πρέπει να προχωρήσουμε, θα πρέπει να προχωρήσουμε γρηγορότερα. Και να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία με τους απεσταλμένους του κουαρτέτου. Α, μια ώρα δεν τα έλεγα μαζί τους στις Βρυξέλλες όταν ήρθανε. Και τους έλεγα τι δυνατότητες βλέπω και του ε, προς να του πείσω πόσο σημαντικό είναι να εκμεταλλευτούμε αυτού του είδου τη συναντήση με του Παλαιστίνιου και δεν με νοιάζει πού θα συναντηθούμε. Δεν πειράζει. Καταλαβαίνω ότι οι Παλαιστίνοι και οι Ισραηλοί πολλέ φορέ ε, αγχώνονται με αυτά τα οποία γίνονται. Οπότε α πάμε στο, στο Ισραήλ να δούμε στην Ιερουσαλήμ τον, τον Εβραίο διομητευτή. Δεν πειράζει. Το θέμα είναι απεσταλμένοι να, να, να, να, να με αυτού που πρέπει, να εξηγούν τι θέσει καλύτερα από ό,τι πριν. Και νομίζω ότι αυτό έχει σημασία για μένα. Μίλησα στον Καρίμ Σαλόμ για την Γάζα και λέγαμε να υπάρχει ένα σημείο, μία γέφυρα, ένα πέρασμα. Και όταν θα γίνει με τις υποδομές, γιατί όταν πήγα στην Γάζα, μιλούσα σε επιχειρήσεις, μιλούσα του νέους και ένα από τα πιο σημαντικά ήταν να υπάρξει τη της οικονομίας, το γρότερο δυνατόν. Είχα συναντηθεί και με τον Ισραηλινό στρατηγό, ο οποίος κάθε φορά ανοίγει το πέρασμα και εκτιμώ τις προσπάθειες που κάνουν και οι Ισραηλινοί. Όμως να εξασφαλίσω ότι το να ξαναρχίσουν οι εξαγωγές αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για το πέρασμα και για την οικονομία. Γιατί αν δεν κινείται η οικονομία ε, δεν γίνεται τίποτα. Και ο Κάριμ Σαλόμ διαπίστωσε και συμφώνησε ότι μπορούμε να κάνουμε τα εξή. Μπορούμε να φτιάξουμε αυτόν τον δρόμο έτσι που να χρησιμοποιείται πιο συχνά. Επίσης, να υπάρχει ο αναγκαίος εξοπλισμός και να, υπάρχουν, να γίνεται πιο γρήγορα αυτό το σκάνι ασφάλεια για να περνάει πιο γρήγορα κόσμο, αλλά και να ε, μάθουν περισσότερο η Παλαιστίνη για το τι, κάνουμε. Θα κοστίσει αυτό πέντε και κάτι εκατομμύρια ευρώ. Θέλουμε μια λύση στη Γάζα και είναι πάντως σημαντικό να γίνουν γρήγορα ό,τι είναι να κάνουμε για να τους βοηθήσουμε. Αυτά είπαμε τον Σαλόμ. Το αυτό το πέρασμα και άλλα περάσματα. Όμως θα πρέπει να δούμε τι συγκεκριμένο μπορούμε να κάνουμε χωρίς να αλλάξει τη βασική μας αρχή. Να ανοίξουν τα περάσματα. Ελεύθερα να κυκλοφορεί ο κόσμος το γρηγορότερο. Κάμπελ. Καλά, να μου επιτίθεστε, αλλά να μην λέτε άλλα για τα περισσότερα από αυτά τα οποία είπατε. Αυτά τα χρήματα δεν είναι για μένα, είναι για αλλού. Για να βοηθήσουμε τα ανθρώπινα τη δημοκρατία, το μέσο της σταθερότητας, η ανάπτυξη κλπ. Σας γνωρίζω και ξέρω και άλλοι από την ομάδα σας. Και όλοι εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο. 100% θέλετε να τους βοηθήσουμε τους Αιγύπτιους και τους Τινήσιους και τους Λίβιους. Και αυτό κάνουμε με αυτά τα χρήματα. Κάνουμε σε όλο τον κόσμο, συνέχεια. 460 ε, εκατομμύρια ευρώ είναι ο προπολογισμό. 135 αντιπροσωπείε χρηματοδοτούμε. Το προσωπικό εδώ, ότι σε όλο τον κόσμο λιγότερο από τα μισά που παίρνει το foreign office. Αν θέλετε να, να με κατηγορήσετε γι' αυτό, αλλά μην μου λέτε ότι έχω δι ευρώ και τα χρησιμοποιώ για ένα πολυτελέ κτίριο. Δεν έχω τέτοια πράγματα. Αυτά έχω και αυτά τώρα εξοδεύω σύμφωνα με τον προπολογισμό που προβλέπετε και προσπαθώ να τα εξοδέψω όσο πιο καλά μπορώ εξυπηρετώντα αυτά που θεωρώ ότι θέλετε κι εσείς να εξυπηρετήσουμε και τα λεφτά τα υπόλοιπα που είπατε πάνε σε αυτούς που τα χρειάζονται. Ε, η Μέση Ανατολή, ναι, αλλάζουν τα πράγματα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και εμείς προσπαθούμε να αλλάξουμε την πλατφόρμα τη οποία λειτουργούμε και προσπαθούμε να δούμε τι δυνατότητε θα έχουμε στην περιοχή. Είτε στο Λίβανο, είτε αλλού και τι μπορεί να γίνει. Βεβαίω ε, αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Αίγυπτο αλλά και στις ε, συζητήσεις... Ε, με τους υπουργού εξωτερικών, μιλάμε συχνά για τις ευκαιρίε που υπάρχουν και που πρέπει να προσφέρονται. Άρα δηλαδή πράγματι ε, μπορούμε να επιφέρουμε κάποιες αλλαγές και θα ήθελα να αναφερθώ και στις σχέσεις που έχουμε. Εγώ εργάζομαι πολύ σκληρά στις σχέσεις με το Ισραήλ και με τους Παλαιστίνιους. Μιλάω με πάρα πολλούς ανθρώπους, με τους ηγέτες και των δύο ε, πλευρών ε, και ιδιωτικά πολλές ώρες και στο πλαίσιο των συναντήσεων και σέβομαι αυτές τις συζητήσεις. Θέλω να σας πω όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται σεβαστή και από τις δύο πλευρές και εγώ θέλω να κρατήσω αυτή τη γραμμή. αυτό είναι και προπόθεση για λύση των δύο κρατών. Μου λένε πράγματα που δεν μου αρέσουν και άλλα που μου αρέσουν. πάντω. πιστεύω ότι και οι δύο σέβονται τη δική μα θέση. Δεν έχουμε περιθωριακό, έχουμε ρεαλιστικό ρόλο. Και ο ρόλο που μπορούμε να διαδραματίσουμε είναι εκείνο που γνωρίζω, που μπορώ να τον προβάλλω. Ε, δεν μπορώ να ε, κάνω αυτό που κάνουν άλλε χώρε. Δεν έχω καν τη δύναμη να το κάνω αυτό. Όμω εκείνο που μπορώ να κάνω είναι να χρησιμοποιήσουμε την πολιτική και οικονομική μα δύναμη έτσι ώστε να στηρίξουμε την ειρηνευτική διαδικασία. Και ε, σε αυτό είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι. Η κυρία Ντότζα είπε ότι απέτυχε πολιτική γειτονία. Όχι, δεν πέτυχε. Βεβαίω θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω. Πριν από αρκετό καιρό είπα ότι πρέπει να θεωρήσουμε την πολιτική αυτή. Τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων απέδειξαν ότι πρέπει να το κάνουμε, να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί, να ε, μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα πράγματα, ευέλικτοι, να αναγνωρίσουμε ότι σε διάφορες χώρες χρειαζόμαστε και διαφοροποιημένη προσέγγιση η οποία πραγματικά θα ωφελήσει τους ε, πολίτες στο τι αυτοί επιθυμούν, ε, στις φιλοδοξίες τους ε, αλλά και στους δικούς μας στόχους. Ειδικοί απεσταλμένοι αυτή τη στιγμή έχουμε ειδικό αποσταλμένο Ο απεσταλμένος στην Τετραμερή είναι ο πολιτικός μας διευθυντής ε, μόλις έχει τελειώσει ο κύριος Σμιτ ε, τη δουλειά του, τότε ε, θα δω τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον, έτσι ώστε πράγματι να είμαστε σωστά εκπροσωπούμενοι στην περιοχή. Και τέλος ε, κύριε Σβόμποντα με ρωτήσετε για τη διέλευση των Ιρανικών σκαφών. Εξ όσων γνωρίζω οι ουρανοί είπαν ότι ήταν μια άσκηση για να ε, αντιμετωπίσουν καλύτερα την πειρατεία στη Σομαλία και γι' αυτό δόθηκε άδεια διέλευσης. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχω. Ε, μόλις τα ακούσαμε ζητήσαμε πληροφορίες έτσι λοιπόν μια τέτοια άσκηση ε, όπως σας είπα για τον λόγο που αναφέρθηκε οι Αιγύπτιοι δεν είχαν λόγο να αρνηθούν τη διάλευση τώρα κατά πόσο αυτό ευσταθεί όχι αυτό είναι άλλο θέμα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και ελπίζω στις απαντήσεις που σας έδωσα να κάλυψα όσο δυνατόν περισσότερα θέματα Πρόεδρος και εμείς σας ευχαριστούμε κυρία Άστον γιατί πράγματι είχατε μια πολύ κουραστική ημέρα ε, δουλέψατε σήμερα πολύ σκληρά εδώ αυτή την αίθουσα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας ε, και μας δώσατε ε, απαντήσεις επί της ουσίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνει η συζήτηση. Θα ξανασυναντηθούμε αύριο. 5η 10 ε, Μαρτίου στις 9 το πρωί μέχρι τη μία το μεσημέρι και πάλι από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Έχει δημοσιευτεί η μερισσία διάταξη και μπορείτε να την βρείτε στις ιστοσελίδα μας. Τελειώσαμε.